Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μετά από ε, ένα τέταρτο καθυστέρηση πάλι, που είναι η συνήθις καθυστέρησή μας. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Πλάς που δέχτηκε να μιλήσει αργότερα, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και θα δώσουμε το λόγο και να παρουσιάσει μέσα σε 20 λεπτά το λόγο της. Τώρα 10 λεπτά, διορθώνει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα που είμαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να σας εξηγήσω κάποια πράγματα που αφορούν τη δομή των γερμανικών αλλά και των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα σας μιλήσω για τη δική μου καταρχήν περίπτωση. Είμαι η ίδια εργαζόμενοι σε μια γεωργική εκμετάλλευση στη Γερμανία και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί να ξαναδούμε τους ορισμούς και αυτά που ακούσαμε επί των οποίων θα συνεχίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας αναφέρω αυτό που διάβασα από τον Άλαν Μάθιους. Όλες οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικογενειακές. Όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι μικρές. Και εδώ μας ενδιαφέρουν κάποιοι πολύ σημαντικοί αριθμοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συνεταιρισμούς, έχουμε κάθε είδους μορφές νομικές ε, οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και μη οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με το μέγεθός τους πολλές φορές τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται η εξοικονόμηση οδηγεί κάποιους γεωργούς στο να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την ε, νομική τους μορφή και υπόσταση. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι σε κάποια κράτη Υπάρχουν συμβατικές σχέσεις. Στην ε, Γερμανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει η λεγόμενη αλληλοβοήθεια, συνεργασία μεταξύ των ε, γεωργών, μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ ε, γειτόνων που μοιράζονται εξοπλισμό, δανείζονται ο ένας από τον άλλον εξοπλισμό, είτε οχήματα, μηχανήματα. Υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασία και υποστήριξη. Γι' αυτό και αυτή η συνεργασία είναι κάτι που πολλές φορές δεν συμπεριλαμβάνεται στις στατιστικές και στα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Πολλά δεν γνωρίζουμε γιατί πολλά ρυθμίζονται με ένα είδος εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών που δεν εγγράφεται και δεν εντοπίζεται από τα στατιστικά στοιχεία. Πολλοί λοιπόν παρουσιάζονται με μεγαλύτερες μορφές ακριβώς επειδή αυτό είναι οικονομικότερο. Είτε παρουσιάζονται με μεγαλύτερες εκτάσεις καθότι αυτό επίσης τους βοηθά να κάνουν οικονομίες κλίμακας. Κάθε είδους οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά και άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβάνονται σε κάποιες κατηγορίες. Θα αναφερθώ εδώ συγκεκριμένα στην Γερμανία όπου έχουμε θέση ήδη από το 1991 22 εκτάρια σαν όριο μεταξύ 20 και 40 εκταρίων είναι οι μεσαίες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για το μέσο μέγεθος τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί το μέσο μέγεθος και αυτό που μας ενδιαφέρει για τις ε, αλλαγές δεν μπορώ να περιοριστώ μόνο στη Γερμανία για να σας δώσω τα στατιστικά στοιχεία. Εγώ προσπάθησα να δω αν θέλετε τα στοιχεία που διαθέτουμε στη Γερμανία. Το 2000 είχαμε 5.000 τρακτέρ τα οποία πουλήθηκαν, αναφέρομαι σε τρακτέρ που έχουν δύναμη, υποδύναμη 74 κιλοβάτ. Πολύ μεγάλα δηλαδή οχήματα, τα οποία ουσιαστικά είναι περίπου το 50% των οχημάτων που πουλήθηκαν στην Γερμανία για το 2000. Τώρα, αν κοιτάξει κανείς τα επόμενα 10 χρόνια, βλέπει ότι στη Γερμανία υπάρχουν 9.000 τρακτέρ 76 κιλοβάρ, δηλαδή το 75% όλων των οχημάτων. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει γενικότερη τάση να αγοράζουν οι Γερμανοί, Γεωργοί όλο και μεγαλύτερα οχήματα, αλλά τελικά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το εργατικό δυναμικό, το κόστος των εργαζομένων, γι' αυτό και προσπαθούν οι Γεωργοί της Γερμανίας να κερδίσουν, να εξοικονομήσουν, να κάνουν οικονομίες κλίμακας αγοράζοντας όλο και μεγαλύτερα οχήματα. Έχουν όμως και μεγαλύτερες εκτάσεις όπως σας είπα γι' αυτό και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και δυνατότητες που τους επιτρέπουν να εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες εκτάσεις με μεγαλύτερα τρακτέρ. Υπάρχουν όμως και πολύ μεγαλύτερα τρακτέρ πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία τα μοιράζονται πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο υποκαθιστούν τους εργαζόμενους. Δεν αυξάνονται δηλαδή οι θέσεις απασχόλησης, αλλά αυξάνεται η υποδύναμη των οχημάτων, των τρακτέρ. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στον τομέα των πουλερικών ή του χείριου ε, κρέατος βλέπουμε παρόμοιες τάσεις. Η Γερμανία εδώ δεν είναι μια μοναδική περίπτωση γιατί βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε από την Eurostat δείχνουν ότι οι εκμεταλλευόμενες ε, δυνατότητες, οι δυνατότητες στις οποίες εκμεταλλεύονται πολλές, ε, πολλά αγροκτήματα είναι μια γενικότερη τάση και μειώνεται ουσιαστικά η έκταση η χρησιμοποιούμενη από το 2003 ως το 2010 οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 2 με 10 εκτάρια μειώθηκαν πάρα πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά εξαγοράστηκαν είτε από πιο μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις πάνω από 100 εκτάρια οι οποίες μεγάλωσαν ακόμα περισσότερα την έκτασή τους. Αυτή είναι μια γενικότερη τάση η οποία φαίνεται, αυξάνεται διαρκώς δηλαδή το μέγεθος και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η τάση και ότι υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Ένα άλλο παράδειγμα πολύ ενδεικτικό είναι ότι, και αυτό το είδαμε από μια μελέτη που είναι στο Γκέτιγκεν, το μέγεθος των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων είναι τελείως διαφορετικό από τη μία περιοχή στην άλλη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και αυτό δεν το λέω μόνο σαν επιστήμον αλλά και σαν αγρότης. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε το λάθος να βλέπουμε τον αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να αυξάνονται χωρίς να κοιτάμε το μέγεθός τους. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε πολλές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης κάποιων οικογενειών. Και αυτό σε πολλές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξειδίκευση, η χρήση νέων τεχνολογιών, η χρήση νέων μηχανημάτων βοηθούν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να περιορίσουμε την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εδώ θα προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία Ράιμερς, η οποία είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε επιπόλαιοι όταν μιλούμε για ορισμό. Μα ζήτησε τι είναι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είναι σίγουρο ότι σήμερα όλες οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμπόδια και θα πρέπει εδώ να δούμε το θέμα του περιβάλλοντος, της οικολογίας, τον ανταγωνισμό που γίνεται σκληρός το λεγόμενο land grabbing, δηλαδή όλο και περισσότερες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο. Οι εκτάσεις, οι επιφάνειες χρησιμοποιούνται όλο, για όλο και περισσότερο για κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αρμοδιότητες πλέον δεν είναι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους και δεν προστατεύονται αν θέλετε οι μικροί ε, γεωργοί, οι μικρές οικογένειες ε, που έχουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έρχονται αν θέλετε επενδυτές ή ε, αρμοδιότητες είναι όλο και περισσότερο αρμοδιότητες, τουλάχιστον στη Γερμανία, περιφερειακές ή των κρατηδίων και βλέπουμε όλο και περισσότερες επιφάνειες να φεύγουν από τη γεωργία και να χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο. Αυτό είναι κρίμα και είναι μια τάση που θα πρέπει να αντιστραφεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επίσης την ανάπτυξη που αποφέρει σε μια περιοχή η ύπαρξη ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ο διεθνής ανταγωνισμός παρόλα αυτά είναι σφοδρός και θα πρέπει να βοηθήσουμε στηρίζοντάς τις, τις μικρές αλλά και μεγάλες ε, οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου όλες οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να είναι οικογενειακές, αλλά όλες οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι μικρές. Υπάρχουν και πολύ μεγάλες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουμε να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο πραγματικό τμήμα της σημερινής απογευματινής συνεδρίασης. Φυσικά αν υπάρχουν ερωτήσεις προς, την, προς τους ομιλητές του πρωινού, όπως προς την κυρία Νταβίδοβα, η οποία είναι ακόμα εδώ, ή προς την κυρία Πλάς, μπορείτε να τις κάνετε. Δεν ξέρω αν η κυρία Χένεση είναι εδώ, αλλά αν έχετε για τις δύο άλλες ομιλήτριες ερωτήσεις, βεβαίως μπορείτε να τις υποβάλλετε πριν προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ ομιλητών. Χρειάζεται ακόμα χρόνο από ό,τι βλέπω για να χωνέψετε τα όσα ακούσατε και να υποβάλλετε ερωτήσεις. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ ομιλητών. Καλούμε βέβαια τους πρωινούς ομιλητές να παραμείνουν στην αίθουσα. Έχουμε τώρα τις διεθνείς προοπτικές. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Λουτσάνο Τζεντόντσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Γεωργίας. Εν συνεχεία, ο κύριος Henri Rouillet d'Orfeuille είναι ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Τσεντόντσε είναι ο πρώτος μας ομιλητής, του δίνουμε το λόγο. <clears throat> Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω ή να προσπαθήσω να παρουσιάσω την άποψη ενός μη κυβερνητικού οργανισμού για τον τρόπο υποστήριξης της οικογενειακής γεωργίας. <clears throat> Λέγομαι Λουτσάνο Τσεντόντζε δουλεύω για μια Ιταλική ΜΚΟ, Τσέφα λέγεται, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 70 ε, Ιταλικές NGOs, μέλη της FOXIV. Μιλάμε για διεθνείς ε, θελοντές ε, που ασχολούνται με την αναπτυξιακή συνεργασία που λειτουργούν και υπάρχουν εδώ και 40 χρόνια για τη δίκαιη και ανάπτυξη. Εκατομμύρια άνθρωποι στο βορρά και στο νότο εμπλέκονται σε δραστηριότητε και project υπέρ της ε, οικονομικής ε, γεωργίας. Θέλω να σας πω τις ε, απόψεις μας για τα εργαλεία που υπάρχουν για την υποστήριξη της οικογενειακής γεωργίας και της διατροφικής ασφάλειας. Στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας, μία ανθρώπινη οικογένεια τροφή για όλους. Ε, με την υποστήριξη της Καριτάς. Η άποψή μας βασίζεται στον κεντρικό ρόλο που έχει ο άνθρωπος και η οικογένεια ε, με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία και ενίσχυση των φυσικών πόρων. Θέλουμε να επιτύχουμε την επιστημιστική ασφάλεια. Το δικαίωμα στην τροφή είναι, είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου θα πρέπει φυσικός πώς και οικονομικός να έχει πρόσβαση σε επαρκή, ικανοποιητική και αποδεκτή τροφή που να έχει παραχτεί με βιώσιμο τρόπο και να λαμβάνει υπόψη και το, το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών. Η βελτίωση του ρόλου των οικογενειών των ε, γεωργών ε, στα πλαίσια της κοινότητάς τους με ειδική έμφαση στο ρόλο των γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε δίπλα στους ε, αγρότες ε, μιλάμε για τα προβλήματά μας, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις ε, και να δημιουργήσουμε πραγματικές εταιρικές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες. Οι γυναίκες και οι νέοι είναι οι βασικοί παίχτες ε, στην αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο για να υπάρξει αλλαγή. Είναι σημαντικό να έχουμε συλλογικές δράσεις που να απορρέουν που να πηγάζουν από την κοινότητα ε, με τη συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας ε, καθώς και τη συμμετοχή βεβαίως οργανωμένων ομάδων ε, γεωργών και νοικοκυριών που μπορούν να διαδώσουν τις αγροοικολογικές καινοτομίες. Η βασική στόχη είναι να ενισχύσουμε τις οικογένειες των γεωργών και τις κοινότητές τους και τις οργανώσεις τους, ούτως ώστε να παίρνουν αποφάση σε τοπικό επίπεδο. Να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για άμεση πρόσβαση και έλεγχο των πόρων και αυτή η προσέγγιση ανταποκρίνεται στην έννοια της α, δημοκρατίας που πρέπει να ισχύει στο χώρο των τροφίμων. Αυτή η προσέγγιση ε, ενσωματώνεται σε ένα πλαίσιο και προκύπτουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές δράσης. Θα πρέπει να υπάρχει ε, η δυνατότητα να καταναλώνουν τα νοικοκυριά ό,τι παράγουν και να μειωθεί η εξάρτησή τους από την εξωτερική παραγωγή. Ε, επίσης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την, τις οργανώσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να προωθηθεί η δημοκρατία και η λογοδοσία. Να υιοθετηθούν αγροοικολογικά συστήματα στη γεωργία λαμβάνοντας υπόψη ε, το συμπληρωματικό ρόλο της ε, οικογενειακής γεωργίας. Εδώ μιλάμε και για την ε, διαχείριση της γης, την δασοκομεία, την διαβίβαση των πολιτιστικών αξιών, διαφοροποίηση πολλαπλά είδη τροφών και ψηλή προστιθέμενη αξία, αύξηση της αφύπνισης, κατάρτιση σε συνεργασία με άλλους τοπικούς εταίρους, ούτως ώστε η οικογένεια των γεωργών να είναι η πραγματική κοινωνική και οικονομική δύναμη της τοπικής ανάπτυξης. Από την εμπειρία της Φόξη, βλέπουμε ότι η αποτελεσματικότητα κάποιων εργαλείων που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής στα νοικοκυριά της υπαίθρου έχουν τα εξής αποτελέσματα. Υποστηρίζουν τις οργανώσεις των παραγωγών, ε, το θέμα της ιδιοκτησίας και χρήσης της γης, ενισχύουν τους τοπικούς πόρους και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στους πόρους, ε, πρόθεση της, της συνεργασίας, των συνεταιρισμών, τις τοπικές οργανώσεις, γίνονται αναγνωρίσιμες, πρόσβαση σε δάνεια και μικροδάνεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο τη οικογενειακή γεωργία για την παραγωγή τη γη και τη διατήρηση. Την παραγωγή, συγγνώμη, τροφίμων και τη διατήρηση τη γη. Επίσης, θα πρέπει ε, να μπορούν οι γεωργοί να καλλιεργούν τις εποχικές, προωθούν εποχικές καλλιέργειες και σοβιές <coughs> και να υπάρχουν κατάλληλοι σπόρ για την, παραγωγή. Επίσης η προώθηση της α, ιδέας του συνεταιρισμού και της οργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να υπάρχει επαρκή στροφή και να υπάρχει να υπάρχουν τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία, θα πρέπει να υπάρχουν και πληροφορίες και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε από πολύ νωρίς στη ζωή για την θρεπτική αξία των τροφίμων. Στο σχολείο, στην οικογένεια, στο σχολείο, ούτως ώστε να καταναλώμε συνειδητά την τροφή μας. Επίσης, οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να μπορούν να αντιστέκονται να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα. Επίσης, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε χαμηλό επίπεδο ε, στις πιο ευπαθείς περιοχές. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα εδάφη, να προωθήσουμε την τη γονιμότητα των εδαφών και τη βιολογική γεωργία. Επίσης, ε, πολιτιστικά, πολιτιστικός πώς η γεωργία έχει υποβαθμιστεί. Είναι σημαντικό να επανακτήσει τη θέση που της πρέπει. Ένα παράδειγμα ενός project όπου όλα τα προηγούμενα αναφέρθηκαν είναι η παραγωγή ε, τοπικού γάλακτος στην Τζόμπε, στην περιοχή Ιρίγκα, στην Τανζανία. Εκεί κατασκευάστηκε ένα εργοστάσιο γάλακτος και κέντρα συλλογής, ούτως ώστε να υπάρχει μια σταθερή αγορά για τους τοπικούς ε, κτηνοτρόφους. Ενεπλάκησαν 850 άτομα και αν βάλουμε και τα μέλη της οικογένειάς 5.000 άτομα ε, είχαν, είχαν 1.500 γελάδες. Τα ζώα τα έλεγχαν οι κτηνοτρόφοι και παρήγαν ε, κατά μέσο όρο 12 λίτρα το κεφάλι, κάθε γελάδα δηλαδή. Τα, το γάλα πήγαινε στο εργοστάσιο, ε, το οποίο είχε δυνατότητα επεξεργασίας 5.000 λίτρα τη μέρα και μεταποίησης 3.500 ε, λίτρα τη μέρα. Η αγορά ε, κρέατος και γιαουρτιού είναι τοπική αγορά και το τυρί επίσης πουλιάται εκεί. Έτσι λοιπόν, μόλις, χάρη στην κατασκευή αυτών των εργοστασίων, το εισόδημα των κτηνοτρόφων για την περίοδο 2010-2012 αυξήθηκε κατά 140%. Επίσης αυξήθηκε και η κατανάλωση γάλακτος στην περιοχή. Μία σημαντική Ιταλική εταιρεία, ε, συνεταιρισμός μάλλον, ε, γαλακτοπαρακοκών υποστήριξαν τους ε, κτηνοτρόφους αυτούς στην Τανζανία. Ε, υπήρξε μια συνεργασία χωρίς να κερδίσουν οι Ιταλοί. Το συμπέρασμα είναι, χάρη στην εμπειρία ε, αυτή διαπιστώσαμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε... για να προωθηθούν πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες πολιτικές ε, που να προωθούν ένα άλλο μοντέλο, πέρα από το άγρο-βιομηχανικό. Ε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αρπαγής της γης να ενισχυθεί η τοπική γεωργία, ε, η τεχνογνωσία, τα... οι δεξιότητες, να δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση της έρευνας, της έρευνας ε, με υποστήριξη της γεωργίας αυτής. Χρειάζονται και άλλες πολιτικές για να προωθήσουμε την τοπική γεωργία και να υποστηρίξουμε τους μικρούς παραγωγούς. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση επίσης στη χρηματοδότηση της οικογενειακής γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Minuta przerwy Πρόεδρος. αν υπάρχει ένα τεχνικό θέμα και θα κάνουμε ένα λεπτάκι διακοπή. Όμω, ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφέρω ότι οι μικρέ εκμεταλλεύσει χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από τι περιφερειακέ αρχέ. Ακριβώ αυτά που είπαμε. Ε, χρειάζεται να ασκηθεί μια περιφερειακή πολιτική για τι μικρέ εκμεταλλεύσει που δεν έχουν μόνο την ε, εμπορική λειτουργία, αλλά έχουν και κοινωνική λειτουργία, κοινωνική διάσταση και εδαφική διάσταση, διότι δεν επηρεάζουν πάρα πολύ την αγορά. Άρα χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Οπότε, για να βοηθήσουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις, δεν κινδυνεύουμε να στρεβλώσουμε τον ανταγωνισμό. Τέλος πάντων, σε αυτό θα επανέλθουμε. Και τώρα να δώσω το λόγο ή στον επόμενο ομιλητή. Okay. Δεν ακούγεται ο μιλητής. Υπάρχει ένα πρόβλημα, φαίνεται. Αχ, μου ζήτησαν, λέει ο κύριος Ορφέκης, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις κοινέ προκλήσεις και για τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τον κόσμο των ε, γεωργών στην Ευρώπη μεταξύ βορρά-νότου δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά όμως κοινά σημεία. Και το πρώτο κοινό σημείο είναι αυτές οι προκλήσεις η Γεωργία παντού στον κόσμο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη, αυτές τις προκλήσεις, δηλαδή να μπορέσει επαρκώ να, να θρέψει 7 δι. και θα πρέπει να υπάρχει κάποιος βιώσιμος, αηφόρος τρόπος διαχείρισης των φυσικών πόρων, αλλά και το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να παράσχει απασχόληση, να αμύψει επίσης με αξιοπρέπεια 40% του παγκοσμίου εργατικού δυναμικού. Και ο Πιζανή είπε το εξή σωστό κάποια στιγμή. Ότι για μπορέσουμε να θρέψουμε τον κόσμο, χρειαζόμαστε τη γεωργία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά για να μπορέσουμε να διχειριστούμε τους φυσικούς πόρους και να μπορέσουμε να... Και για τέλος να μπορέσουμε να, να δώσουμε αυτή την αξιοπρεπή ε, αμοιβή στου ε, στους εργαζομένους του πλανήτη χρειαζόμαστε τη γεωργία όλου του πλανήτη. Οπότε θα ήταν καταστροφικό να αποκλείσουμε κάποια περιοχή, κάποια μορφή γεωργίας. Επομένως χρειαζόμαστε τη γεωργία, κάθε μορφή γεωργίας. Και χρειάζεται επίσης να δούμε την πολλαπλή, τις πολλαπλές λειτουργίες των ε, γεωργικών ένα Άλλο κοινό σημείο είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει μια τριπλή επανάσταση παντού. Χρειάζεται μια εντατικοποίηση της παραγωγής. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΦΑΟ, θα χρειαστούμε πάνω από 70% παραγωγής και αυτό θα γίνει με εκτατικοποίηση αλλά και με εντατικοποίηση. Δεύτερον, όσον αφορά τη διαχείριση των ε, φυσικών πηγών και για το περιβάλλον, χρειάζεται να γίνει κάποιο είδους ε, η αγροτοοικολογική επανάσταση, μια επανάσταση και στα μέσα στους μεθόδους παραγωγής. Επίσης χρειάζεται να γίνει μια επανάσταση, ούτως ώστε να μην αποκλείεται κανείς από την απασχόληση στη γεωργία και θα επανέλθουμε σε αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Η τρίτη ε, προσέγγιση το κοινό σημείο κάθε γεωργίας είναι ότι χρειάζεται κρατική πολιτική και επίσης ε, ρύθμιση διεθνής. Πρόσβαση στις αγροτικές γέες. χρειάζεται να εξασφαλιστεί η χρήση των αγροτικών γεών και από πλευράς κυριότητος, αλλά τουλάχιστον στην Γαλλία οι παραγωγοί θέλουν να υπάρχει κάποια συνέχεια, κάποια σταθερότητα, να μην υπάρχει ένα καθεστώς που κάθε φορά θα πρέπει κάθε γενιά να αγοράζει, να ιδιοποιείται τη γεωργική γη. Επίσης, χρειάζονται κάποιες τιμές που να κρίνονται από σταθερότητα. Αλλιώς, δεν μπορεί να γίνει υπάρχει ρύθμιση. Δεν θα πρέπει να έχουμε ανισορροπίες. Χρειάζονται επομένω κάποιες αμοιβέ σταθερές βασικό αυτό και για επενδύσεις και για καινοτομία. Μιλάμε για επιδοτήσει, αλλά αυτό δεν είναι κρατική επένδυση. Πρόκειται για επένδυση των παραγωγών ακόμα και στη φτωχή Αφρική. Και εκεί οι περισσότερε επενδύσει προχωρούν από του ίδιου του παραγωγού. Αλλά για να υπάρξουν ε, επενδύσει θα πρέπει το, το, το, το εισόδημα των παραγών να είναι επαρκές. Επίσης χρειάζεται πρόσβαση σε κάποιο είδους πιστώσει, σε δανειοδότηση που να συνάδει προς την γεωργική παραγωγή. 3% ετησίως είναι αυτά τα δάνεια. Αλλά στις περισσότερες χώρες εξαφανίζονται τα αγροτικά δάνεια. Πολλές φορές φτάνουμε σε τέτοιου είδους ε, ε, επιτόκια του 3-4% κατά μήνα πολλές φορές, το οποίο είναι καταχρηστικό. Επίσης μια άλλη πολιτική είναι το ότι χρειάζονται κάποιες κρατικές υποδομές. Δρόμοι, έρευνα, Χρειάζονται επομένω υποδομέ και επίση χρειάζεται πρόσβαση σε συμβατέ προσαρμοσμένε τεχνολογίε. Χρειάζεται ένα σύστημα που να διακρίνεται από καινοτομία. Χρειάζεται, να, όπως έγινε στην Αφρική, να υπάρξει κάποια τέτοια προσαρμογή και συνοδευτικά μέτρα γιατί όταν δεν είναι αξιόχρη η παραγωγή σε κάποιες χώρες δεν έρχεται να βοηθήσει ο δυτικό τομέα. Άρα εδώ πέρα μπαίνει ο λόγος των ε, οργανώσεων των παραγωγών που βοηθούν αυτές τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αυτό γίνεται και από διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς χώρες. οι εισοδές δεν είναι μόνο για τις ε, οικονομικές επιχειρήσεις. Ας πούμε η Βραζιλία έχει κάνει ε, μεγάλες προόδους παράλληλα και με, με τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και στις οικογενειακές. Και ε, σε πολλά μέτρα. Πρώτα-πρώτα καταπολέμησαν την ε, εξαθλίωση στην Ήπεθρο Έχουν μια τέτοια πολιτική και δεν στοχεύουν ειδικά την Γεωργία, αλλά προσπάθησαν να βοηθήσουν τους πιο φτωχούς. Και επίσης πολιτικές χωροταξίες προσπάθησαν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους μη προνομιούχους και έτσι βοήθησαν και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν και μετά και πιο ειδικέ ε, πολιτικές στην ε, Βραζιλία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά τα, τα δάνεια. Κάθε μέρα έχουμε 45 εκατομμύρια γεύματα στα σχολεία. Και υποχωρεί αγορά 30% στις οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις από αυτά τα σχολεία. Και οπότε έχουμε μια τέτοια διάσταση περιβαλλοντική, κοινωνική, χωροταξική Τώρα κάτι άλλο που θα να σας ε, σχολιάσω είναι το ζήτημα του ορισμού. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τα σύνορα. Όπως και να ορίσουμε την οικογενική γεωργία, θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα κριτήρια για να δώσουμε σωστό ορισμό. Είναι θέμα αν είναι ορεινή περιοχή, ε, μέγεθος, τέλος πάντων κάποια άλλα κριτήρια, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό είναι η οικογενειακή γεωργία. Γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχουν κάποιες εκμεταλλεύσεις που χρειάζονται άλλες που δεν χρειάζονται να καλυφθούν. Και χρειάζεται κρατική πολιτική και Έχουμε κάποιες σοβαρές απειλές όσον αφορά την κερδοσκοπία, το κεφάλαιο προς τις γεωργικές γέες και η αντίδραση είναι το να αναδείξουν το γεγονό ότι σχεδόν η πάντως όλη γεωργία είναι οικογενειακή γεωργία. Σε αντίθεση με το μοντέλο το οποίο έχει τόσο πολύ ευνοηθεί παντού. Οπότε το θέμα δεν είναι η επιχείρηση ενός παραγωγού, αλλά δεν υπάρχει ένα άλλο μοντέλο ως προς να βρει τη διαχείριση και έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές ομοιότητες παντού και ίδιους στόχους στον κόσμο, αλλά υπάρχει μια σημαντική ανισορροπία ανάλογα με την περιοχή, την περιφέρεια, ε, το είδος της ε, κρατικής πολιτικής που ασκείται χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες μερικές παρατηρήσεις ότι εξορισμού η γεωργία είναι μια δραστηριότητα που γίνεται σε διαφορετικό, διαφορετικά περιβάλλοντα ε, πολλές δυσκολίες υπάρχουν κάποιες, υπάρχει κάποιο είδους φυσικής στρέβλωσης Οπότε ανταγωνίζονται μεταξύ τους πολύ διαφορετικά είδη γεωργίες. Επίσης, στο Νότο είναι οι πιο φτωχή γεωργία και ενώ εδώ την ε, Αφρική, ε, στην Ασία, γιατί εκεί δεν υπάρχει κάποιο οικονομική υποστήριξη, ενώ στον Βορρά υπάρχει οικονομική βοήθεια. Δηλαδή εκεί στο Νότο ε, υπάρχει λίγη καθόλου βοήθεια. Ε, ενισχύσει ε, δασμοί. Ανατολική Αφρική είναι πολύ φτωχή και είναι επομένω η περιοχή η πιο ανοιχτή, η πιο ευάλωτη στον κόσμο. Και όταν έχουμε κάνει μια τέτοια γεωργία που δεν έχει υποστήριξη, τότε δεν είναι δυνατόν να κερδίσουμε την παγκόσμια μάχη που δίνουμε για τη γεωργία. Αν θέλουμε επομένω να επιβιώσει η Γεωργία παντού σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν τι πιο μεγάλες δυσκολίες και που είναι πιο ευάλωτε στον ανταγωνισμό. Επίσης, ε, η διεκδίκηση των Αφρικανών ε, εκφράζεται με κάποια οργάνωση που υπάρχει και λέει ότι εκεί που πετύχατε εσείς ε, το ίδιο ζητάμε και εμείς και μας το αρνείστε. Οπότε το πρόβλημα ακριβώ το θέμα ότι δεν μπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισμό οι Αφρικανοί. Επίση να σταθούμε σε ένα άλλο σημείο την πρόκληση που αφορά την απασχόληση που είναι ο τρίτος άξονας αυτής της τριπλής επανάσταση. Και εδώ θέλω να σταθούμε διότι Νομίζω ότι σχεδόν 100% συμφωνούμε γιατί ξέρουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει εντατικοποίηση της παραγωγής και αυτή η αγροοικολογία ότι χρειάζεται και έχει όμως και αυτή την πτυχή που αφορά την απασχόληση και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ βορρά και νότου. το γεωργοδημογραφικό επίπεδο που διαφέρει. 65% των ε, ανθρώπων στην Αφρική ασχολούνται με αυτό, 50-55% στην ε, Ασία και στον ΩΣΑ κάτω από 5%, 3% στην Γαλλία, 1,5% στη ΣΥΠΑ και 40% είναι ο όρος ο παγκόσμιος και από το 60 μέχρι το 3% ε, ήταν μια εξέλιξη που κράτησε 150 χρόνια στην Ευρώπη, στη Γαλλία τέλο πάντων. Οπότε, για να δούμε τώρα ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση. Ένα δις είναι το, το πρόβλημα της απασχόλησης. Αυτό χρειάζεται να βρούμε 1,1 δις Θέσουν στην απασχόληση και τι θα γίνει μέχρι το 2050, αν θα αυξηθεί ή όχι το, το, πρόβλημα. Σχεδόν, σχεδόν τελειώνω. Για να δούμε τι θα θα δημιουργήσουμε θέση απασχόληση. μεταξύ 15 και 60 ετών είναι αυτοί, αυτά τα 900 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης που λείπουν. Και για να δούμε την απολογή δημογραφικής, όλοι συμφωνούν ότι θα έχουμε μέχρι τότε 2 ε, εκατομμύρια περισσότερους, 2 δις. Και αυτοί θα είναι σε, σε ηλικία ενεργή, οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς δεν θα καταστραφούν οι θέσεις απασχόλησης στην Γεωργία. Και αν πάμε μόνο σε αυτό το, το, μοντέλο του 3% αντί για το 40% βλέπουμε ότι θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια, 2,6 δις που θα καταλήξουν την Γεωργία και όλοι αυτοί πρόκειται να ψάχνουν δουλειά. Άρα, έχουμε αυτούς που σήμερα δεν έχουν δουλειά Έχουμε επομένω 3,8 δις θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαμε να καλύψουμε. Εάν δεν καταστραφούν θέσεις απασχόλησης, επομένω συμπερασματικά για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο, αυτό το μοντέλο του 3% του πληθυσμού ασχολείται με την Γεωργία είναι ένα πρόβλημα σχεδόν άλυτο, τουλάχιστον για Αφρική και Ασία. Το δε θέμα του, της περιθωριοποίησης των ε, χωρικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές συνέπειες. Και μόνο εάν δεν περιθωρούμε κανέναν έχουμε τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τριπλή πρόκληση που σας ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτών των διεθνών πτυχών που αφορά, αφορούν την οικογενειακή γεωργία, το πώς έχουν τα πράγματα εκτός Ευρώπης, γιατί βλέπουμε πόσο μεγάλη ποικιλία υπάρχει. Και τώρα σας προτείνω να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις, να δώσουμε τις απαντήσεις και έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Κύριο Άγνιο, έχει ζητήσει τον ε, λόγο με τα Βοητσέφσκη και κατόπιν Καπούλα Σάντος. Άγνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όλους το λέω αυτό. Υπάρχουν δύο δυναμικές δύο τρόποι με τους οποίους προχωρεί, προχωρούν οι γεωργοί, η γεωργία στο Ηνωμένο Βασιλείο, εξάρτητα από τα μέτρα της ΚΑΠ ή της μεταρρυθμίσης της ΚΑΠ. Καταρχάς, η κάθετη ολοκλήρωση, όπου τα σούπερ μάρκετ θέλουν απόλυτη χνηλασιμότητα και ο οικογενειακός, ο μικρός α, γεωργός, τελικά θυσιάζει όντως την ανεξαρτησία του, αλλά του εγγυώνται ένα, μια λογική τιμή για τα προϊόντα του, εφόσον χρησιμοποιεί τα στοιχεία παραγωγής που το, που το σούπερ μάρκετ του, υποδεικνύει. Γιατί θέλει το σούπερ μάρκετ απόλυτη χνηλασιμότητα και θέλει να ξέρει από πού προέρχονται τα στοιχεία παραγωγής. Μπορεί λοιπόν με αυτό το σενάριο να επιβιώσει ο μικρός οικογενειακός γεωργός, αλλά δεν είναι τόσο ανεξάρτητος όσο θα ήθελε. Είναι κακό αυτό κατά τους ομιλητές. Α, ίσως είναι καλό, γιατί κρατάει μακριά τις εισαγωγές. Γιατί τα εισαγωγές, εάν κρατήσει αυτό το μοντέλο το σούπερ μάρκετ, οι εισαγωγές δεν μπορεί να εξασφαλίσουν απόλυτη χνηλασιμότητα. Θα θυμάστε, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, γιατί ας πούμε όταν έγινε πέρυσι το, το σκάνδαλο, με το αλογίσιο κρέας, θα θυμάστε ότι λέγανε που πουλάνε, ότι πουλάνε ας πούμε βόλιο κρέας και πουλούσαν αλογίσιο. Γι' αυτό χρειάζεται η χνηλασιμότητα. Ας πούμε, επίσης οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι ε, συνειδητοποίησαν ότι ο κίνδυνος εκτροφής γουρουνιών ε, είναι μεγάλος. Οπότε τι κάνανε, στην πραγματικότητα ε, νίκιαζαν το χειροστάσιο και δάνειζαν ε, το άχυρο κτλ. Στην πραγματικότητα ε, δεν ήταν πια κτηνοτρόφοι, απλώς νίκιαζαν την υποδομή τους και μίστοναν το εργατικό τους δυναμικό. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, υπάρχει μια αντίσταση από τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Εάν, ας πούμε, ένας ε, γεωργός θέλει χίλιες αγελάδες ε, γαλακτοπαραγωγής, χρειάζεται άδειε. Και συχνά ε, οι υπόλοιποι εκεί στην κοινότητα δεν το θέλουν κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν, ας πούμε, ε, οι αγελάδε έχουν όλε τι ανέσει, τη μοντέρνα τεχνολογία, αν υπάρχει κτηνοτρόφος μόνιμα που πηγαίνει εκεί σε αυτέ τι μεγάλε εγκαταστάσει. Ακόμα κι αν η κοπριά, α πούμε, ε, την επεξεργαστούν ούτω ώστε να μην μυρίζει η περιοχή κτλ. Πολύ υγιεινέ όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, αποτελεσματικές κτλ. Και, και πολύ φιλικές για τους γύρω. Αλλά αυτός ο αριθμός ζώων σε ένα μέρος ε, συγκεντρωμένο ενοχλεί τον κόσμο στη χώρα μου. Προσπαθούν λοιπόν να μην επιτρέψουν να δοθούν τέτοιε άδειε για τέτοιε εγκαταστάσει. Μπορεί να πει κάτι λοιπόν από το κάποιο ομιλητή από το πάνελ για αυτέ τι τάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές, γιατί ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Το θέμα των ε, οικογενειακών ε, εκμεταλλεύσεων είναι κάτι που πραγματικά μας ενδιαφέρει στην Πολωνία παραδείγματος χάρη, στο σύνταγμά μας. Υπάρχει μία διάταξη που αναφέρεται ακριβώς στην οικογενειακή γεωργία και επί πολλά χρόνια υπήρχε η πίεση να αλλάξει αυτό και να υπάρξει μία νομική πράξη που δίνει πραγματική προτεραιότητα και προτίμηση στις ε, οικογένειες που ενεργοποιούνται στην γεωργία. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ένα πρόβλημα αν θέλουμε να στηρίξουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στην οικογενειακή γεωργία, διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά στρέβλωση του ανταγωνισμού και αντιτίθεται στους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να εκφράσουμε εδώ την προτίμησή μας για την οικογενειακή γεωργία που να συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν έχουμε όλο και μεγαλύτερα αγροκτήματα, μεγάλες ε, βιομηχανικού τύπου γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τόσο εύκολα, αν θέλετε, την οικογενειακή γεωργία, ενώ αυτό είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας, κάτι που πρέπει να παραμείνει ζωντανό στο μέλλον. Το δεύτερο σημείο είναι η γη η οποία είναι διαθέσιμη για τους γεωργούς. Η κατάσταση διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Εμείς όταν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε μία δωδεκαετή περίοδο κατά την οποία ξένοι δεν μπορούν να αγοράσουν εκτάσεις στη χώρα μας. Όμως αυτή η μεταβατική περίοδος δυστυχώς τελειώνει και βεβαίως η κατάσταση από τη μια χώρα στην άλλη είναι τελείως διαφορετική. Στη Γαλλία παραδείγματο χάρη θεωρητικά μόνο ε, θεωρητικά οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει γη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στην πράξη αποκλειστικά και μόνο Γάλλοι αγρότες ε, διαθέτουν την γη. Και στη Γερμανία η κατάσταση είναι διαφορετική. Στην ε, Πολωνία όμως δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν είναι ίσως θέμα υπηκότητας γιατί αν κάποιος γεωργός από μία ξένη χώρα θέλει να αγοράσει γη στην Πολωνία, αυτό θα έπρεπε να επιτρέπεται. Εμείς φοβούμαστε όμως ότι θα αυξηθούν οι ανισότητες και ότι οι πιο φτωχές ε, γεωργικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί περισσότερο το θέμα. Δεν είναι καθαρά δικό μας πολωνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Οι διαφορές δυστυχώς δεν εξαλείφονται τόσο εύκολα και οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης συνεχίζουν να διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές. Εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 10 χρόνια. Οι διαφορές όμως συνεχίζουν. Και αυτό που δυστυχώς επιδεινώνει την κατάσταση είναι ένα πολύ άδικο σύστημα εξισορρόπησης και άμεσων πληρωμών. Όσον αφορά τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εγώ συμφωνώ ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζονται από κοινοτικά κονδύλια. Τι γεωργία θέλουμε, φυσική, βιώσιμη, παραδοσιακή ή με γενετικά τροποποιημένες διαδικασίες και οργανισμούς. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε και να επιδοτούμε τέτοιου είδους γεωργία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ήταν ερώτηση αυτή, αυτή ήταν παρουσίαση. Ο κύριος Καπούλα Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, ομιλητές για τις παρουσιάσεις. Εγώ είμαι από μια χώρα με μεγάλη ιστορική παράδοση στην οικογενειακή γεωργία, ήδη από την ε, κατάργηση των δικαιωμάτων ε, του πρωτότοκου γιου από το 19ο αιώνα ήδη οι πολύτεκνες ε, γεωργικές οικογένειες παρέμεναν στη γεωργία με τον κατακαιρματισμό της γης και με πολύ πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εγώ σαν εισηγητής της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής Γνωρίζω πολύ καλά τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για τις μικρές και τις πολύ μικρές γεωργικές ε, εκμεταλλεύσεις και σε μια περίοδο κρίσης, σαν και αυτή που γνωρίζει σήμερα η Ευρώπη, βλέπουμε οικογένειες στη γεωργία που ουσιαστικά εργάζονται στη γεωργία αλλά και σε άλλους τομείς. Έχουν δηλαδή και άλλες προσοδοφόρες δραστηριότητες για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους γιατί η γεωργία δεν αρκεί για να επιβιώσει μια οικογένεια. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ περήφανος για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στον τομέα αυτό και πιστεύω ότι παρόλο που υπήρξαν μεγάλες αντιστάσεις από βουλευτές που δεν ήθελαν να στηρίξουν την οικογενειακή γεωργία. Παρ' όλα αυτά εμείς καταφέραμε να περάσει το καθεστώς αγρότη, να υπάρξει ένα καθεστώς ανακατανομής, να εισάγουμε κατόφλι όσον αφορά την στήριξη και βεβαίως τα μέτρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος για εκμεταλλεύσεις κάτω από 10 εκτάρια. Όλα αυτά βεβαίως δεν αρκούν. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την κυρία Πλάς και μου φαίνεται ότι άκουσα μία επίκριση σε σχέση με την αναδιάρθρωση κάποιων εκμεταλλεύσεων. Η αλήθεια είναι ότι πολλές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αν δεν είχαν και άλλες δραστηριότητες εκτός από τη γεωργία, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Οι μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια μόνο από το γεωργικό τους εισόδημα. Πολλές φορές υποχρεώνονται οι γεωργοί να εγκαταλείψουν τη γεωργία. Τα 25 τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία, στον τομέα του γάλατος, παραδείγματος χάρη, είχαμε 80.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην χρονιά που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε 7.000. 7.000 που παράγουν το διπλάσιο από αυτές που είχαμε με 80.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό οφείλεται όχι μόνο στον αριθμό των ζώων, των αγελάδων για κάθε αγρόκτημα, αλλά και από την απόδοση και το μέγεθος αυτών των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κυρία Πλάς, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλήσατε για την συγκέντρωση πολλών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι το αρνητικό. Αν όμως δεν είναι βιώσιμες αυτές οι μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αν δεν αρκεί το εισόδημά τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, γιατί είστε κατά της αναδιάρθρωσης και από τι επίπεδο, τι μέγεθος και πέρα δέχεστε την αναδιάρθρωση. Μπορείτε να μου απαντήσετε κυρία Πλάση. Γιάρ Καρινόφσκι είναι οι τελευταίοι δύο ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω σημειώσει εδώ ότι οτιδήποτε είναι κακό για την ανάπτυξη είναι κακό και για την οικονομική ανάπτυξη, ότι είναι κακό όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου της γεωργίας. Ε, το θέμα εδώ είναι να δούμε τι ακριβώς ε, είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη, για δυναμική εξέλιξη στην γεωργία, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα μεγάλου μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βιομηχανοποιημένη γεωργία. Βεβαίως, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν πολλές φορές ε, και πολλά πλέον εκτίματα. Η βιωσιμότητά τους βασίζεται, παραδείγματος χάνει στην ευελιξία μιας οικογενειακής εργασίας. Οι οικογένειες ε, πολλές φορές μπορούν να θεωρηθούν πιο βιώσιμες, έχουν μια μελλοντική προοπτική, καθότι υπάρχει μια νέα γενιά, άρα καινοτομία, άρα χρήση νέων τεχνολογιών. Το θέμα τώρα είναι, και αυτό το ακούσαμε και το πρωί, πώς ορίζουμε την οικογενειακή εκμετάλλευση. Πώς ορίζουμε τις διάφορες κατηγορίες ως προς το μέγεθος. Σήμερα ξέρουμε ότι ο τομέας της γεωργίας επίσης γνωρίζει μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Εξού και βλέπουμε πάρα πολύ λίγους νέους να στρέφονται προς αυτό το τομέα. Το θέμα των μεγάλων ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αγοράζουν, εξαγοράζουν τις ε, μικρές. Αυτό είναι το ένα. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω, γιατί η πρώτη μου ερώτηση ήταν τι είναι κακό σε αυτή την ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά η δεύτερη ερώτησή μου είναι ότι ναι, είναι κάτι θετικό η οικογενειακή γεωργία. Μπορούμε όμως να τη βάλουμε στο κέντρο, στην καρδιά μιας πολιτικής, ε, μιας στρατηγικής. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την οικογενειακή γεωργία. Μια οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση έχει δικαίωμα να ζήσει από την δραστηριότητά της. Έχει επίσης δικαίωμα να υποστηριχθεί με εξοπλισμό, με χρηματοδότηση και έχει το δικαίωμα να ε, στηριχθεί όσον αφορά την ανάπτυξή της, την εξέλιξή της. Δεν έχω, αν θέλετε, πολιτικές λύσεις να προτείνω, γι' αυτό και θα ήθελα να σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Καλινόσκη. Τρία την θέλω να σας αναφέρω πρώτα φορά τις διαρθρωτικές ε, αλλαγές που συνέβησαν δεκαετία του 90. Ε, στην Πολωνία είχαμε 800.000 ε, που ασχολούνται με την ε, ε, γαλακτοκομία και την σχετική μεταποίηση. Τώρα έχουμε 180.000 τέτοιου γεωργού που ασχολούνται με την κτηνοτρόφους α πούμε, την γαλακτοκομεία. Πάντως νομίζω ότι αυτή η αλλαγή ήταν θετική εξέλιξη. Θα συνεχιστεί πάντως να αλλάζει το τοπίο στην Πολωνία Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προ το συμφέρον μα, σα τα λέω όλα αυτά από πλευρά Πολωνία ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο τη Δυτική Ευρώπης, από και από κοινωνική πλευρά, όπως ακριβώς προαναφέρατε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης. Επίσης, ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η κυρία Πλάς ότι θα πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στη στατιστική όταν ε, ε, ασκούμε την πολιτική μας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα πρέπει κανείς να μελετήσει βαθύτερα το τι γίνεται. Στην Πολωνία έχουμε 1.400.000 Πολωνών οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσει για επιδοτήσεις. Αυτό συνάδει προς τα στατιστικά που ισχύουν ε, μπαίνει αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Ε, γιατί το 1 τρίτον αυτών που ζητούν τις επιδοτήσεις δεν είναι πραγματικοί ε, καλλιεργητές. Απλώς ζητούν επιδοτήσεις διότι είναι κύριοι αγροτικών γεών που κάποτε χρησιμοποιείται για γεωργία ή κτηνοτροφία, αλλά δεν χρησιμοποιείται πια κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει στην Πολωνία το, τι θα, το θέμα του τι θα γίνει με την Γεωργία όταν σταματήσει η μεταβατική περίοδος για τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τη χώρα μας. Αλλά να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένα, κατόπιν το, τον όσων είπε ο κ. Βοητσεχόφσκι πριν, εάν εξετάσετε το τι τι, τι λύσεις δώσαν οι Δανείοι, οι Γάλλοι πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιες νομικές ε, παρεμβάσεις στο σύστημα της Πολωνίας όσον αφορά ας πούμε το άνω όριο, το maximum του πόσο μπορεί το κράτος να παρεμβαίνει να παρεμβαίνει στη δομή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οπότε έχουμε αυτό το φόβο του τι θα γίνει τότε μετά τη μεταβγή περίοδο. Πάντως θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά, γιατί άλλων υπάρχουν ρυθμίσεις και άλλων εφαρμόζονται σωστά. Πάντως θα συνεχιστούν οι αλλαγές στη χώρα μας. Ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανείς άλλος να δει το λόγο. Α, όχι, όχι. Να, κάποιος δει το λόγο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο είπε ο συνάδελφος για την ε, Πολωνία. Λέει ο κύριος Άγνιο. Ε, λέω ότι όλοι αυτοί ζητούν επιδοτήσεις χωρίς όμως να ασκούν γεωργική δραστηριότητα. Είναι κύριο όμω της γεωργική γεία. Τι γίνεται όμως εκεί. Τι συμβαίνει σε αυτές τις ε, γεωργικέ γεία που κατέχουν αυτά τα πρόσωπα. Ίσως ε, δεν αναφέρθηκε με τόση ακρίβεια συνάδελφος, μήπως ασκείται η δραστηριότητα, αλλά όχι τόσο τόσο, τόσο, τόσο, τόσο εντατικά. Δεν ξέρω αυτό πώς ξέφυγε από τη μετάφραση. Καλινόφσκι. Ναι, ναι, ναι, ασκείται κάποια δραστηριότητα γεωργική, όπως είπε σωστά ο πρόεδρος. Αλλά αυτή η δραστηριότητα εξελίσσεται, ασκείται με τέτοιο τρόπο που ας πούμε ότι δεν, δεν, επίσημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η γεωργία. Τώρα θα να απαντήσουν όσο πιο σύντομα γίνεται οι προσκεκλημένοι μα από το πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τα παραδείγματα που αναφέρατε. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές τα στατιστικά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις και πόσο μεγάλο είναι το φάσμα τελικά το, της γεωργίας και των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Δεν θέλω ούτε να επικρίνω, ούτε να αξιολογήσω εδώ, αλλά πραγματικά Νομίζω ότι όταν μιλάμε για μια οικογενειακή εκμετάλλευση δεν αναφερόμαστε μόνο σε μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, είπατε να δώσουμε την άποψή μας για το πώς βλέπουμε την εξέλιξη. Αν κοιτάξει κανείς άλλες αγορές, όπως τη Νέα Ζηλανδία, θα διαπιστώσει ότι η η απελευθέρωση της αγοράς έδωσε τέτοιες νέες δυνατότητες, ο ανταγωνισμός παραδείγματος χάρη, που σήμερα μπορούμε να αναρωτηθούμε αν είμαστε σε θέση να επιβιώσουμε στην Ευρώπη σε έναν τέτοιο ανταγωνισμό. Ναι, ναι. Έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια αγορά, υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει βιωσιμότητα θα επιβιώσουν τελικά οι περισσότερες επιχειρήσεις οικογενειακές. Εσείς αναφερθήκατε στην περίπτωση της Πορτογαλίας και δώσατε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρόκειται για ταχύτατες μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές. Η κυρία Νταβίντοβα μίλασε σήμερα για την γύρανση του πληθυσμού, παραδείγματος χάρη. Ίσως ε, αυτό συνέβη και σε εσά. Δηλαδή, η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να οφείλεται στο ότι υπήρχε λιγότερη λιγότερο ενδιαφέρον από τις νέες γενιές ότι οι περισσότεροι αγρότες ήταν ηλικιωμένοι και δεν υπήρξε διαδοχή. Ίσως αυτό οφείλεται και ο περιορισμός ε, του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δεν θέλω να το αξιολογήσω, δεν θέλω να πω αν είναι κάτι καλό ή κάτι κακό, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι αν δεν μπορεί να αντισταθεί και να ανταποκριθεί, να ανταπεξέλθει μια γεωργική εκμετάλλευση στον ανταγωνισμό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι είτε εξαγοράζεται από κάποια άλλη επιχείρηση, είτε εξαφανίζεται. Δεν θέλω να πω ότι μόνο οι μεγάλες θα επιβιώσουν. Το βιώσιμο μοντέλο δεν οφείλεται μόνο στο μέγεθος. Πρέπει πραγματικά να δούμε πού υπάρχουν προκλήσεις, πού υπάρχει η δυνατότητα να ανταπεξέλθει κάποιο στον ανταγωνισμό και σίγουρα, σίγουρα μετά θα πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές μας. Ευχαριστώ. Να απαντήσω και σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Κάποια από αυτά που είπατε για την οικογενειακή γεωργία στην Ευρώπη μοιάζουν, μας παραπέμπουν ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί γεωργοί στην Αφρική. Ένα από τα προβλήματα των Αφρικανών ε, γεωργών, μικρών γεωργών, είναι να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Ε, επομένως πρέπει να υπάρξει μια καλή οργάνωση των δομών. Πιστεύουμε ότι για τοπικά προϊόντα υπάρχει τοπική αγορά. Όταν μιλήσαμε για την υποστήριξη στους γεωργούς στην Αφρική ή στην Ασία ή στην Κεντρική Αμερική ή στην Νότια Αμερική, δεν νομίζουμε ότι εννοούμε εδώ την υποστήριξη για τις εξαγωγές. Το βασικό είναι να υπάρξει αυτάρκε σε τοπικό επίπεδο, να έχουν πρόσβαση οι γείτονε στα τοπικά προϊόντα της ε, εκμετάλλευσης και πρόσβαση των ε, προϊόντων στις τοπικές αγορές. Προτείνουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και μετά τις εμπειρίες που είχαμε στην Ιταλία και στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια εντοπίσαμε διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Φερρυπίν η Αφρική είναι αντίστοιχα με αυτά που αντιμετώπιζε η Γεωργία στην Ευρώπη τη δεκαετία του 50 ή του 60. Θέματα ε, οργανωτικά, θέματα πρόσβασης σε πιστώσεις, θέματα πρόσβασης στις αγορές. θέματα προσόντων και δεξιοτήτων. Και τέλος, το θέμα της ε, κοινωνικής αξίας της γεωργίας. Αυτό που συμβαίνει ας πούμε στην Κένια, εκεί δουλεύουμε εμείς και την ξέρουμε την περιοχή. Οι γεωργοί επενδύουν χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτοί που το κάνουν αυτό δεν έχουμε τα εργατικά χέρια για την εκμετάλλευσή τους. Τα παιδιά τους δηλαδή που τα σπουδάζουν, κυρίως τα αγόρια, όταν πάρουν το παραμικρό δίπλωμα, εξαφανίζονται από τη γεωργία. Γιατί δεν θεωρείται αξιοπρεπής δουλειά. Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, να αλλάξουμε το μοντέλο γεωργίας, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γεωργία, που, που τη βλέπουν τη γεωργία. Αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία, Φερρυπίν. Τι βλέπουμε να συμβαίνει. Υπάρχει μία σχολή γεωργικών σπουδών και υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητέ να σπουδάσουν εκεί. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ανιχνευσιμότητας και ποιότητα των προϊόντων από την Αφρική. Όχι πια, όχι σήμερα. Εδώ και ένα κάποιο χρονικό διάστημα έχει εκλείψει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά όχι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο τελευταίο μιλήτη να συνοψίσει. Πρώτη παρατήρηση του Άγγλου ομιλητή. Είναι παγκοσμιοποιημένο το επιστηστικό μας σύστημα. Έχουμε μαζική παραγωγή, ε, μαζική διανομή, κατανάλωση, μαζική κατανάλωση αν θέλετε. Εξάλλου και ο ΠΟΗ ΠΟΕ αυτό το μοντέλο προωθεί και αυτό το σύστημα το επιστηστικό έχει τα πλεονεκτήματά του. Καταρχάς έχει τις τιμές. Με συνεχεία. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, εξασφαλίζει την πρόσβαση και σε ό,τι αφορά την υγειονομική ασφάλεια. Υπάρχουν λιγότερα νεκροί ε, λόγω διατροφής από ό,τι θα είχαμε σε ένα σύστημα κατακαιρματισμένο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αρνητικά ε, εξωτερικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία και παράμετροι. Καταστρέφουμε φυσικούς πόρους, ε, μολύνουμε την υδροφόρο ορίζοντα λόγω κάποιων μοντέλων γεωργίας που προωθούμε και κοινωνικά υπάρχουν προβλήματα συγκέντρωσης, επομένως αποκλεισμού κάποιων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που υπάρχει παντού στον κόσμο, νομίζω, είναι ότι δημιουργούνται ε, εδαφοποιημένα ε, πιστιστικά συστήματα που έχουν μια άλλη λογική, που συνδέουν τη γεωργία με τον τόπο όπου γίνεται, που δημιουργούν ένα πλαίσιο σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή ε, φέρουν κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή, που δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην απασχόληση και στο περιβάλλον, γιατί όλα αυτά γίνονται σε μικρότερη, κλίματα, μικρότερη κλίμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική όπου έχουμε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις. Ε, οι μεσαίες ε, εκμεταλλεύσεις ε, επλήγησαν από την κρίση. Όχι οι μικρές οι οποίες αν δεν είναι εντελώς απομονωμένες μπορούν να πάνε προς αυτό το μοντέλο που σας ανέφερα και μακριά τις αγορές. Είναι σημαντικό αυτό το εδαφικό σύστημα να το βοηθήσουμε. Είναι και προς όφελος κάποιων από, τον, από τους καταναλωτές. Ε, σημαίνει ποιοτικά προϊόντα, αν υπάρχει η χνηλασιμότητα των προϊόντων, έχουμε μπροστά μας τον παραγωγό, έχουμε αυτή την επιλογή. Εγώ μελέτησα τις α, περιφερειακές πολιτικές 22 περιφέρειες της Γαλλίας. Ε, όλες είναι υπέρ αυτού του μοντέλου. Υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές υπέρ αυτού του μοντέλου. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα για τις υπόλοιπες. Το δεύτερο ερώτημα, σημαντικό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο δίκαιο για να υπερασπιστούμε τις ε, οικογενικές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Χρειάζονται πάντως α, ε, πολιτικές. Το 1960 στη Γαλλία έγινε μεγάλη μεταρρύθμιση γεωργική που έδωσε εξουσία στις οργανώσεις παραγωγών Είχαμε το τον κύριο Πιζάνη υπουργό τότε. Είχαμε δύο ε, νοικοκυριά αναγεωργική εκμετάλλευση. Και έτσι ε, η έγκυα πολιτική ε, βασίστηκε σε αυτό το μοντέλο. Ε, υπήρξε μια εποπτεία της ε, έγκυας αγοράς, αποφύγαμε τις πολιτικές όπου μεγαλώνει εκμεταλλεύσεις άμετρα. δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό το μοντέλο στους, στα παιδιά των γεωργών. είναι οι εκμεταλλεύσεις, αλλά ε, όλα αυτά έγιναν βαθμία. Επίσης, το μέγεθος των ε, εκμεταλλεύσεων, ε, ο αριθμός των εργαζομένων, αυτό το θέμα δεν είναι μόνο γεωργικής φύσεως. Είναι ένα θέμα που συνδέεται με την αγορά εργασίας. Αν έχετε όλα τα στοιχεία για να εντάξετε στον χώρο εργασία αυτού που φεύγουν από τη γεωργία, υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε γεωργίε 3%, 3% α πούμε. Ε, η διαρθρωτική ανεργία εμφανίστηκε στη Γαλλία το 70%. Συγγνώμη, το δεκαετία του 70. Έγινε αυτή η έξοδος ε, των εργατικών χεριών από τη Γεωργία σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη εκβιομηχάνηση. Οπότε απορροφήθηκαν αλλού. Αν έχουμε, τώρα όμως που έχουμε 3-4 μόνιμα ανέργους, όταν έχουμε διαρθρωτική ανεργία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να εξαλειφθούν οι μικροί γεωργοί για να μπουν στη μαύρη τρύπα. δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Επίσης, ε, στη Γεωργία υπάρχουν πολύ μικρές οικονομίες κλίμακος. Ε, σίγουρα καλύτερα να έχεις 3.000 ε, εκτάρια παρά 3, αλλά για την κοινότητα δεν έχει σημασία. Δεν έχουν σημασία οι μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις. Ε, σίγουρα για την κοινότητα, αν κάνουμε τον υπολογισμό, ε, του εθνικού συμφέροντος και της παραγωγής, ίσως καλύτερα να έχουμε 3.000 εκμεταλλεύσεις από ένα εκτάριο την καθεμία, ειδικά αν υπάρχει πρόβλημα εργασίας. Ειδικά από τη στιγμή που μπορούμε να φτιάξουμε συνεταιρισμούς, να ομαδοποιήσουμε τον κόσμο κτλ. Οικονομίες κλίμακας τότε δεν θα υπάρχουν βέβαια. Αλλά μπορούμε να έχουμε με εντατική παραγωγή μικρές εκμεταλλεύσεις. Λίγες οικονομίες κλίμακας βέβαια. Φυσικά η ιδέα ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί με 1000 εκτάρια παρά με 10 ισχύει στην αρένα πηγική ή στη μεγάλη βιομηχανία αλλά δεν ισχύει στη γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος για το, την τελευταία παρέμβαση, για αυτό το κομμάτι της ακροασής μας. Θα διακόψουμε για ένα λεπτό για να αλλάξουν τα μέλη του πάνελ. Και τώρα, προχωρούμε στο δεύτερο τμήμα στη συνέχεια που αφορά την συμμετοχή το πιστεύω τέλο πάντων των ίδιων των ε, Γιώργων. Πώς βλέπουν αυτά για τα οποία συζητήσαμε οι ίδιοι οι ε, αγρότες. Έχουμε τον κύριο Στέφη από την Τσεχία, τον κύριο, την κυρία Σβάρτσμαν από την Αυστρία και τον κύριο Άντεμς από την Λετωνία. Καλώς ορίσατε. Πρόεδρος, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι και ξεκινούμε. Για άλλη μια φορά, καλώ ορίσατε. όπω προείπαμε, αυτό είναι το πιο κατάλληλο συμπέρασμα ή τέλο πάντων πιο κατάλληλο κλείσιμο. Διότι θα δώσουμε πρώτα πρώτα το λόγο στον κύριο Στέφλ από την ε, Τσεχία. Ξέρουμε ότι έχετε ιδιόμορφε ε, συνθήκες να ε, αντιμετωπίσετε. Γιατί περάσατε από τον μετασχηματισμό της χώρας σα από το καθεστώς ε, του κομμουνισμού στο σημερινό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Γιάν Στέφιλ. Έχω 16 εκτάρια και ασχολούμαι με τη βιολογική γεωργία και έχω άλλα 35 για συμβατική γεωργία. Και με βοηθάει η γυναίκα μου στη διαχείριση και κρατάει και τα βιβλία, κάνει τα λογιστικά. Έχουμε από το 2011 το γιο που βοηθάει, αλλά έχουμε επομένω ε, και πολλά μοσχάρια και επίσης ε, έχουμε και παραγωγή αμύλου. Πατάτες, επίσης. Ε, επίσης έχουμε και βοσκοτόπι, αλλά έχουμε και φερζοαλωνιστική μηχανή. Ανήκουμε σε μια οργάνωση με 2.500 παραγωγών και επίσης ανήκουμε και στον φορέα, τη συνεταιρισμού, τέλο πάντων, των ε, κτηνοτρόφων βοήου κρέατος. Αλλά ασχολούμεθα και με εκτροφή αλόγων και οπότε ανήκουμε και σε, εκείνη την, σε εκείνο τον φορέα. Θεωρούμε ότι το καλύτερο μοντέλο είναι αυτό το οποίο ακολουθούμε εμείς, δηλαδή η παραδοσιακή γεωργία και έτσι θα έχουμε βιώσιμη γεωργία και ε, βιώσιμη τέλος πάντων ε, κτηνοτροφία και αηφόρο. Επίσης ε, θεωρούμε ότι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις των χιλίων εκταρίων και άνω ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το κέρδος από ότι εμείς. Θεωρούμε ότι εμείς θα μεταλαμπαδεύσουμε αυτού του είδους την παράδοση στις επερχόμενες γενναίες. Το 2014 ε, είπαμε ότι είναι η χρονιά των, ε, των γυναικών εκμεταλλεύσεων, οπότε και εμείς θα γιορτάσουμε το, τους ανθρώπους της ε, στη χώρα μας. Επίσης είναι το οικουμενικό έτος της ε, φαμίλιας και νομίζουμε ότι ε, αυτό που μας βοηθάει είναι ότι μία γενιά παραδίδει την εκμετάλλευση στην επόμενη. Θεωρούμε ότι βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση του περιβάλλοντος και το σοφή του περιβάλλοντος. Είναι μια γεωργία που κρατάει αιώνες, έχει, έχουμε φυσικούς δεσμούς με το περιβάλλον και επίσης ε, έτσι ε, προλαμβάνουμε την υποτίμηση, την απαξίωση της γης. Επίσης ε, έχουμε την παραγωγή και ε, τα προϊόντα πάνε από την φάρμα στην, ε, ε, στην αγορά, έχουμε φυσική εκτροφή ζώων και επομένως αποτελούμε το σύνδεσμο μεταξύ Πέθρο και, της, και των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο. Έχουμε ένα διτό σύστημα στην Τσεχία. Συνδυάζουμε δύο διαφορετικά στοιχεία και έχουμε πρώτα πρώτα τις, τους μεγάλους συνεταιρισμούς οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα που ε, έχουν μέλη γεωργούς οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία σε μισθωμένα εδάφη. Επίσης, έχουμε και στην Ένωση Παραγωγών τις οικογενειακές εμμεταλλεύσεις που από το 99 και μετά ε, διεκδικούν πίσω τις γης που τους είχαν αφαιρεθεί από το προηγούμενο καθεστώς. Βλέπετε τώρα αυτές τις διαφάνειες. Κοιτάξτε, φαίνεται εδώ πέρα η εξέλιξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Βλέπετε σε ποια κατάσταση ήταν όταν οι συνεταιρισμοί επέστρεψαν τις ε, ε, αφαιρεθήσεις ε, μεταλλεύσεις τους κυρίους τους και βλέπετε τι έγινε, τι εξέλιξη υπήρχε μέσα σε 10 ή 20 χρόνια. Το από το 99 λοιπόν, ξεκίνησαν από το 0 αυτοί οι γεωργοί και τώρα έχουν προοπτικές ε, για το μέλλον. Βλέπετε εδώ σε αυτές τις φωτογραφίες πώς ήταν σαν αυτή δεκαετία του 90 και πώς είναι σήμερα. Οπότε θα πρέπει να σας πω εν κατακλείδη ότι συνήθως σε αυτές τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ε, δυστυχώς τους αρνείται το Υπουργείο μας την οικονομική υποστήριξη. Μιλώ όχι μόνο για τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, μιλώ για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Μέχρι τα 30 ή 50 εκτάρια. Ανάλογα με το, την τοποθεσία. Και επομένω είναι πάρα πολύ θλιβερό το ότι το Υπουργείο Γεωργίας, τέλο πάντων οι αρχές αρνούνται κάθε χρηματοδότηση, κάθε ενίσχυση όπως ε, προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλουν να υποστηρίξουν τις εκμεταλλεύσεις γενικά ανεξαρτήτως μεγέθους. Και για, πάντως, για τη φύση και για την κοινωνία αντίθετα οι γονείς εκμεταλλεύσεις αποτελούν σημείο στήριξης. Σας ευχαριστώ. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σφάρτσμαν από την Αυστρία. Έχετε το λόγο, κυρία Σουάρτσμαν. geschätzte και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας μπορούμε να πάρουμε το λόγο εδώ στο Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά έχει συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την οικογενειακή γεωργία κάτι που είναι αυτονόητο αν θέλετε στο παρελθόν και στην παράδοση είναι για μας μια λύση για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύουμε πραγματικά ότι εδώ όλοι αυτοί που συνεισφέρουν στην οικονομία και στην πολιτική με αυτόν τον τρόπο, συνεισφέροντας με την προσωπική τους και οικογενειακή τους ε, εργασία με οικολογικό τρόπο και προστατεύοντας το περιβάλλον. Βλέπουμε ότι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η γεωργία σήμερα που πάσχει από έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε πολλούς τομείς θα πρέπει να εγγυηθούμε και τη βιωσιμότητα και την ιχνηλασιμότητα και την ποικιλομορφία. Και πολλοί είναι αυτοί που σήμερα θεωρούν ότι στον τοπικό πληθυσμό, στους γεωργούς της Ευρώπης υπάρχουν σήμερα οικογένειες οι οποίες εργάζονται στον τομέα αυτό και αυτό έχει μια προστιθέμενη αξία. Εμείς, η οικογένειά μου και εγώ θέλω να δείτε πού ζούμε. Και είμαι σίγουρη ότι κοντά στην λίμνη της ε, Κωνσταντας και κοντά στην περιοχή που ζούμε, με μια μικρή επιφάνεια, 11,5 εκτάρια με αγελάδες, γαλακτοφόρες και πουλερικά, και διάφορες άλλες δραστηριότητες ε, το καλοκαίρι. Ζούμε σε ορεινή περιοχή και με πέντε άλλες οικογένειες έχουμε και μία θερινή δραστηριότητα, δηλαδή στο πιο ορεινό σημείο της περιοχής μας εκτρέφουμε και γαλακτοφόρες ε, αγελάδες, παράγουμε τυρί με πολύ συγκεκριμένη αν θέλετε ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη και πουλούμε τα προϊόντα μας αυτά, τα τυριά που είναι πάρα πολύ ωραία για το πρωινό, αυτό είναι μια παράδοση της περιοχής μας, κατευθείαν στους καταναλωτές. Στην περιοχή μας, επαναλαμβάνω, οι δραστηριότητες είναι πολλές και διαφορετικές. Όσον αφορά τώρα τη δικιά μας γεωργική εκμετάλλευση. Υπάρχουν πάνω από 130 διαφορετικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μικρές, μεσές, 19 εκτάρια και μόνο 5% αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ξεπερνούν τα 100 εκτάρια. Στην Αυστρία, κατά μέσο όρο 5,2 άτομα ζουν και εργάζονται στην κάθε γεωργική εκμετάλλευση και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών, περίπου το 19% είναι οικογενειακές, 36% αυτών έχουν επικεφαλής μια γυναίκα. Το 70% της καλλιεργήσιμης γης ουσιαστικά ανήκουν στις ορεινές περιοχές στην Αυστρία. Πρόκειται για μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες εργάζονται παραδοσιακά και φυσικά πρόκειται για λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, ορεινές περιοχές, τις οποίες ουσιαστικά λειτουργούν πολλές πολλά διαφορετικά είδη γεωργίας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Και έχουμε δομές οι οποίες είναι διαφανείς, εύκολο κατανόητες, ποικιλομορφία των προϊόντων, καθώς και αυτό που ονομάζουμε σε μας η διατήρηση του τοπίου. Το τοπίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ψυχαγωγία, ο τουρισμός είναι σημαντικά για την περιοχή μας και γι' αυτό και η χρησιμοποίηση εξοπλισμού και μηχανημάτων ακόμα και στις πιο εντατικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις γίνεται με πολύ λογικό και προσεγμένο τρόπο γιατί για μας η διατήρηση του τοπίου του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κάνουμε λοιπόν όπως σας είπα πωλήσει επιτόπου στο αγρόκτημα ε, οικολογικό τουρισμό, αγροτουρισμό, κάτι που μας βοηθάει για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της περιοχής μας αλλά και τους τουρίστες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό δεν είναι το κόστος, δεν είναι η τιμή αλλά πραγματικά η ποιότητα. Θέλουμε να δείξουμε στους τουρίστες και στους πολίτες της περιοχής μας ότι αυτή η ποικιλομορφία, αυτή η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να διατηρήσει τις οικογένειες επιτόπου με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε επίσης να αναπτύξουμε αυτή τη γεωργία, αυτή την ποιοτική γεωργία σε αυτές τις ορεινές περιοχές η οποία βεβαίως έχει και πολύ θετικές κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή. Στήριξη για τους πολίτες των περιοχών αυτών που με αυτόν τον τρόπο παραμένουν στις περιοχές μας καθότι ο τρόπος επιβίωσης τους υποστηρίζεται από την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εμείς πραγματικά στηρίξαμε αυτή την ανάπτυξη της υπαίθρου προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε με κατάρτιση, με προγράμματα τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις πιο μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν βιώσιμες και να βοηθήσουν τις οικογένειες αυτές με δυναμικό τρόπο να παραμείνουν στις ε, οικογενειακές τους εκμεταλλεύσεις. Προσπαθούμε επίσης να δώσουμε νέες δυνατότητες, κάτι που πολλές φορές ε, οφείλεται και στην οικογενειακή δομή. Η οικογένεια πρέπει να τύχει στήριξης. Σε εθνικό επίπεδο στην Αυστρία έχουμε προγράμματα στήριξης της οικογένειας, της ε, διαδοχής από τη νέα γενιά. Εγώ θέλω και επιθυμώ να παραδώσω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου μία ε, επιχείρηση η οποία να είναι καλύτερη από αυτή που παρέλαβα. Και αυτό βεβαίως δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική βιωσιμότητα αλλά και στην ποιότητα αυτού το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε. Επαναλαμβάνω ότι η ύπεθρο, το τοπίο, η ποιότητα της ζωής, η βιωσιμότητα αυτών των εκμεταλλεύσεων είναι πραγματικά οι εγγυήσει για να παραμείνουν επιτόπου οι πολίτες των περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει αυτές τι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα σταθεροποιητικό παράγοντα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πολιτική στήριξη της οικογένειας, ακριβώς επειδή παίζει και έναν οικονομικό αλλά και κοινωνικό ρόλο. Οι δημόσιες ε, πολιτικές στήριξης, οι παροχές μπορούν να βοηθήσουν στο να ενδυναμωθεί αυτός ο πυλώνας. Οι οικονομικές, γεωργικές εκμεταλλεύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και θα πρέπει να τις στηρίξουμε και όχι να τις αποδυναμώσουμε. Στην Ευρώπη αυτό το επιτυχημένο μοντέλο θα πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο στην βιώσιμη οικονομία και στην διατήρηση της υπαίθρου και του τοπίου των περιοχών μας. Ευχαριστώ, Λέω Φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους ακροατές θα θέλουν να πάρουν τα στοιχεία σας για να έρθουν στην περιοχή σας να περάσουν τις διακοπές τους. Στην πλαγιά σας, στην εκμετάλλευσή σας. Και τώρα ο κ. Άνταμς από την Λετωνία. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Γεια σας, λέγομαι Κάσπαρ Άνταμς, είμαι από τη Λετωνία. Είμαι 28 χρονών. Νέο. εντάξει, ανάλογα και πώ το βλέπει κανεί και πώς χρονών είναι. δουλεύω στην ε, Ήπεθρο, παλιότερα δούλεψα με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, έχουμε μια μικρή εκμετάλλευση και βλέπετε από το βιογραφικό μου ποιο είναι το μέγεθος μετακλευσή μα. Οι γονεί μου ξεκίνησαν την γεωργία το 1994. Τώρα έχουμε 300 κεφάλια βοηθών, έχουμε 600 ε, εκτάρια, τα 300 είναι δικά μας και τα 300 τα πνικιάζουμε. 600 εκτάρια μπορεί να μοιάζουν πολλά, αλλά αν τα συγκρίνουμε με το πόσα εκτάρια έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε άλλες χώρες, δεν είναι και τόσα πολλά. Στη Λετωνία υπάρχει πολύ ανεκμετάλλευτη γη που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε για γεωργία και αρχίζουμε λίγο-λίγο να την καλλιεργούμε, την καθαρίζουμε, την ξεχερσώνουμε, βγάζουμε τους τάμνους και επεκτηνόμαστε. Επομένως, το δυναμικό της γεωργίας στη Λετωνία είναι μεγάλο σε σχέση με τις ειρηνητικμένες χώρες όπως η Γερμανία, Φερπίν οι γονεί μου είναι Και έχουμε διαφορετικές απόψεις στην ε, εκμετάλλευσή μας. Εγώ έχω φιλοδοξίες και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Το 2010 λοιπόν δημιούργησα με την βοήθεια των γονιών μου μία δημοπρασία, ένα χώρο δημοπρασίας για τα βοηδή. Είναι η μοναδική δημοπρασία που γίνεται για βοηδή στη Λετωνία. Θα μιλήσω λίγο αυτό αργότερα. Θέλω να σας πω όμως ότι και ο παππούς μου ήταν αγρότης από το 1954 και μετά. Ε, ασχολήθηκε με, τον, ε, με τα κτηνιατρικά. Ε, έφερε, με, εισήγε ζώα από τη Γαλλία. Εγώ από παιδί ε, συμμετείχα. Συμμετείχα σε αποφάσεις, στις συνεδριάσεις, στη συζητήση για το πώς θα αναπτύξουμε την ε, φάρμα μας και νομίζω ότι έμαθα από τα λάθη που κάνει παλιή. Βλέπετε και από το φυλάδιο που σας, μίλησα, που σας μοίρασα ότι πιστεύω πως όλοι μπορούν να βρουν τη θέση τους στην, Ήπειρο, στην Ήπεθρο. Ε, οι νέοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην Ήπεθρο. προτιμούν ανάμεσα στα δύο να πάνε στην πόλη να δουλέψουν. Αν του θέσει το ερώτημα η η πολη Πιστεύω ότι για να είναι μια πετυχημένη γενιά, από γενιά φάρμα από γενιά σε γενιά, θα πρέπει να βρεις λύσει λύσεις και μάλιστα να συμφωνήσουν οι γονείς με τα παιδιά. Α, ε, δεν μπορεί από μόνος να κάνεις κάτι χωρίς τη βοήθεια των γονιών σου. Φυσικά υπάρχουν πολλοί νέοι γεωργοί κτηνοτρόφοι που ξεκινάνε το μηδέν και τότε είναι πολύ σημαντικό να κάπου να βρουν μια στήριξη. Πιστεύω ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν οργανώσεις που βοηθούν ε, με την ανταλλαγή εμπειριών, ε, με τις επισκέψεις που οργανώνουν, με την ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών, και με τη συνεργασία γενικά, η οποία επεκτείνεται από χρονιά σε χρονιά τους γεωργούς. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι μπορώ ε, να δουλέψω σήμερα για να αφήσω μια καλύτερη κατάσταση στα παιδιά μου. Και η καλύτερη κατάσταση θα εξασφαλιστεί και από την ε, δημοπρασία που οργάνωσα. Εκεί ε, πουλούνται τα βοηθή στη μεγαλύτερη, στην ψηλότερη δυνατή τιμή. Κάποια νούμερα για την αγορά βοήου στην Λετωνία. 20 ε, αγελάδες έχει μέση φάρμα στη Λετωνία. το ζωικό κεφάλαιο είναι 744, 50 εκτάρια είναι το μέσο, η μέση έκταση μιας ε, φάρμας. Φυσικά υπάρχουν και φάρμες που έχουν 1.000, 2.000 εκτάρια. Αλλά Εντάξει, συμβαίνει αυτό στη Δανία. Ε, συμβαίνει αυτό στην Λετωνία, αλλά στη Δανία, ας πούμε, μου είπε ένας φίλος από τη Δανία ότι σπάνια ε, υπάρχουν τόσο μεγάλες φάρμες. Μάλιστα, μία μόνο έχει 2.000 εκτάρια. Το 90% των ε, βοηδών εξάγεται στην Ευρώπη. Εμείς δεν τρώμε και πολύ βόλιο ε, και η οικονομική κατάσταση δεν είναι πολύ καλή τώρα για να καταναλώνεις βόλιο το οποίο είναι τόσο ακριβό. Επομένως, εξάγουμε τα ζώα μας για τις ε, δημοπρασίες ζώων. Εγώ αυτό το φτιάξα από το μηδέν. Φυσικά δεν είναι νέο για την Ευρώπη αυτό, αλλά για τη βαλτική περιοχή είναι κάτι το πρωτοφανέ, το καινοτόμο για το εμπόριο των βοηδών. Έχουμε μια οργάνωση όπου συμμετέχουν 700 κτηνοτρόφοι και συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις. Δεν είναι, η οργάνωση που έχουμε δεν είναι συνεταιρισμός ως προς τη νομική της μορφή. Δημιουργήσαμε στο παρελθόν κάποιες, ε, κάποιους συνεταιρισμούς οι οποίοι απέτυχαν, εξαφανίστηκαν και δεν αναλάμβανε τις ευθύνες τους. Γι' αυτό διάλεξα άλλη νομική μορφή. Εγώ οργανώνω τις ε, δημοπρασίες και όσοι κτηνοτρόφοι θέλουν να συμμετάσχουν, συμμετέχουν. Μέσα σε τέσσερα χρόνια έγινε πολύ δημοφιλής η δημοπρασία αυτή και έτσι και Λιθουανοί και Εστονοί συμμετέχουν. Φυσικά δεν μπορεί να φέρει κανεί τα βοηθή του από πολύ πιο μακριά. Ε, επίσης, στη Λετωνία εμείς α, εξυγχρονίζουμε τις φάρμες μας, αυτό που προνομήσαμε από τη Σοβιετική εποχή. Επίσης, οι μεγάλες φάρμες, ε, ή μάλλον οι φάρμες που θέλουν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο, χρειάζονται και τα οικονομικά μέσα για να αναπτυχθούν. Οι μικρές ε, γεωργίες εκμεταλλεύσεις έχουν μικρότερη πρόσβαση στην πίστοση και επομένως δεν μπορούν να αναπτυχθούν όσο θα ήθελαν. Σε, σε, αν τις εγκρίνουμε με τις μεγαλύτερες, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο. Επομένως ο κόσμος προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες φάρμες, μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Επίσης η δημοπρασία βοήθησε τις μικρές εκμεταλλεύσεις, γιατί μέχρι τότε, αν ήθελε κάποιο να πουλήσει τι αγελάδε του, ε, χρειάζονταν και λεφτά για να οργανώσει την πώληση. Ενώ τώρα υπάρχει ήδη μία δομή και δεν έχει σημασία αν θα πουλήσει μία ή περισσότερες, ε, υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όμως στη Γεωργία και για να αρχίσουμε να επιλύουμε τα προβλήματα αυτά, πιστεύω ότι ένας τρόπος είναι να προσελκύσουμε νέους, μορφωμένους ανθρώπους στη Γεωργία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την εκπαίδευση. Πέρσι υπήρχε ένα project από την Ευρωπαϊκή Ένωση για νέους γεωργούς και στην... το αποτέλεσμα ήταν ότι στην κτηνοτροφία ενδιαφέρθηκαν 50 νέοι Λετονοί. Δηλαδή, αποφυτώντα από τα πανεπιστήμια αυτοί 50 νέοι, αποφάσισαν να αναλάβουν την ε, γεωργική εκμετάλλευση των γονιών του και να δουλέψουν εκεί. Κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειδικά στη Λετωνία, είναι το γεγονός ότι η Ήπεθρος δεν έχει μόνο την ε, κοινωνική διάσταση, γιατί φυσικά η γεωργοί όταν αγοράζουν πράγματα δίνουν και δουλειά σε άλλους. Ή, ας πούμε πουλάνε τα προϊόντα τους για την παραγωγή ζωοτροφών. Η ύπεθρος πρέπει να γίνει και πιο ελκυστική ως τοπίο. Η τελευταία απειλή που είδαμε για την Ήπεθρο είναι η σταθμή βιοαερίου. Η ιδέα είναι πολύ καλή από μόνη της, αλλά πιστεύω ότι είναι καλή μόνο όταν εμπλέκονται και οι γεωργοί. Όταν υπάρχει, όταν υπάρχει ας πούμε, μια φάρμα, ας πούμε μια φάρμα γαλακτοκομικών προϊόντων και χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα για να παράγουν βιοαέριο. Και εν συνεχεία χρησιμοποιούν αυτό το αέριο για το γενικό καλό. Το ίδιο πράγμα δεν είναι καλό όταν τις ε, δουλειές αυτές, δημιουργία σταθμών ε, βιοαερίων, τις κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Φτιάχνουν, ας πούμε, ένα σταθμό βιοαερίου στο κέντρο μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Ενός αγρού. Και σε μια ακτίνα 50 χιλιόμετρων είναι πολύ δύσκολο να αγοράσει κανείς γη, γιατί οι τιμές είναι να νοικιάσει ε, γιατί τα νίκια ανέβηκαν εκθετικά, οι τιμές των πρώτων υλών εκτοξεύθηκαν στα, ύψη. Στην περιοχή που ζω εγώ πριν από δύο χρόνια υπήρχε ένα project για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος σταθμός. Αλλά οι τοπικές αρχές είπαν stop. Φυσικά υπάρχουν περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τέτοιοι σταθμοί και που δεν τους, και δεν ανήκουν στους γεωργούς και τότε η κατάσταση για τους γεωργούς είναι αρκετά δύσκολη. Συμπερασματικά. Η γη είναι ως είναι. Δεν μεγαλώνει, δεν πολλαπλασιάζεται, δεν αλλάζει αυτό, δεν το επηρεάζει. Αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στα όσα μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη γη για γεωργικούς σκοπούς. Και θα πρέπει η γεωργία να είναι μορφωμένη. Και το πιο σημαντικό είναι να προσελκύσουμε στην Ήπεθρο νέους. Νέους, νέους. Ε, Ευχαριστώ πολύ <laughs> για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Και τώρα να είστε πολύ σύντομοι, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση στις 5. Σας παρακαλώ πολύ, σύντομα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν, στον ομιλητή από την Τσεχία μιλήσατε για τις οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις και την υποτίμηση της γης, τη μείωση της τιμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε πρόκειται για μικρή γεωργική εκμετάλλευση, είτε για μεγάλη εντατική καλλιέργεια, γιατί εσείς μας μιλήσατε για μείωση της τιμής. Μήπως ήταν λάθος αυτό που άκουσα, η μετάφραση. Επίσης, όταν αναφέρεστε στις πληρωμές, Μπορείτε να μου αποσαφηνίσετε τι ακριβώς εννοούσατε στην κυρία από την Αυστρία. Συγχαρητήρια. Μας μιλάτε για την δική σας εκμετάλλευση 11,5 εκτάρια και λέτε ότι μπορείτε να ζήσετε. Μπράβο. Επίσης ε, είπατε ότι κάνετε και άμεσες πωλήσεις μέσω ενός δικτύου λιανικού εμπορίου πουλάτε κατευθείαν τα προϊόντα σας. Μπράβο σας, θεωρώ ότι πραγματικά αυτό είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Τέλος, είστε ένας νέος από την Λετωνία και πραγματικά αυτά που κάνετε είναι εξαιρετικά. Ίσως ε, θα φτάσετε και μέχρι την συνταξιοδότηση σε κάποια χρόνια. Μιλήσατε για το για το βιοαέριο αέριο και αναφερθήκατε σε κάποιες εγκαταστάσεις Δεν κατάλαβα ακριβώς όμως τι κάνετε με αυτό το αέριο. Το εμφιαλώνετε. Το στέλνετε. το στο εθνικό δίκτυο, το πουλάτε στο εθνικό δίκτυο. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γέγκλε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη τις παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε και αυτή για την Αυστρία. Ουσιαστικά είδαμε τρεις προσωπικότητες διαφορετικές, οι οποίες εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι μακριά από τη δική σας ε, περιοχή και πραγματικά ουσιαστικά αυτά που ακούμε εδώ μοιάζουν πολύ με αυτά που γνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό σαν ε, κοινωνία, σαν νοοτροπία και σαν υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους τομείς να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η διαφορά μεταξύ μιας οικογενειακής, αν θέλετε, ε, επιχείρησης και μιας μη οικογενειακής είναι η ευθύνη. Και ακριβώς αυτό είπατε, αυτό που σας συνδέει, αυτό που σας δένει με την επιχείρησή σας είναι αν θα μπορέσετε να το μεταβιβάσετε στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι κάτι που για μας πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία, να είναι σημαντικό. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις κατεξουσιοδότηξη πράξεις και το θέμα ήταν παρόμοιο. Ο καθένας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει σε αυτό το γραφειοκρατικό άχθος. Και δώσατε πολύ καλά παραδείγματα. Είπατε πολύ συγκεκριμένα ότι κανείς στην ε, επιχείρησή σας δεν μπορεί να κάνει τη διοικητική, τη γραφειοκρατική εργασία. Μόνο εσείς. Άρα αυτή θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Και πραγματικά αυτό που συζητήσαμε σήμερα το πρωί και ελπίζω και η Ελιζάμπετ θα συμφωνήσει εδώ μαζί μου, το δικό σας παράδειγμα, τα δικά σας παραδείγματα δίνουν μια απάντηση σε αυτό που λέγαμε σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις, λοιπόν. Πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, έπρεπε να μας δώσετε μία συμβουλή και να εκφράσετε μία επιθυμία. Τι θα λέγατε, τι σας φαίνεται το πιο καυτό αν θέλετε. Κοιτάξτε, δεν σας έχω ξανακούσει έτσι, αλλά και εγώ πραγματικά θα ήθελα να σας πω ότι την ίδια ερώτηση με τον Πίτερ ήθελα να κάνω και εγώ, να σας ρωτήσω εσάς ε, τι θα θέλατε να μας πείτε. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί Έχουμε τόσο λίγο χρόνο να περάσουμε μαζί σας. Εσείς είστε οι εμπειρογνώμονες, εσείς γνωρίζετε καλύτερα το τι συμβαίνει στη γεωργία στην Ευρώπη. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε το πρωί από τους καθηγητές και από τους ερευνητές στον τομέα αυτό, αλλά εσείς, η δική σας γνώμη είναι η πιο σημαντική. Πραγματικά θέλω να σας ακούσω κι εγώ τι περιμένετε από εμά. Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις ήταν πολύ θετικές για σας. Ο κύριος Άγνη είναι ο μόνος που έκανε πραγματική ερώτηση. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε. Έχετε ένα λεπτό ο καθένας. Zur e- Πρώτη ερώτηση. 11,5 εκτάρια σε ορεινή περιοχή. Ελπίζω και αυτό να το ακούσατε. Ναι, μπορούμε να επιβιώσουμε γιατί πραγματικά η πολυμορφία των δραστηριοτήτων μας είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Δεν μπορώ εδώ να σας μιλήσω για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι πολύ διαφορετικές οι δομές όμως στην περιοχή μας. Και δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε παραπάνω λόγω της μορφής της περιοχής. Θέλουμε να παραμείνει ζωντανή η περιοχή μας, ζωντανό και όμορφο το τοπίο μας, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία, για όλη την περιοχή. Και γι' αυτό και βάζουμε στο επίκεντρο της ε, δραστηριότητάς μας τον άνθρωπο. Βεβαίως χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη, έτσι ώστε με χαρά και ευχαρίστηση να συνεχίσουμε να είμαστε δραστήριοι και να εργαζόμαστε στην περιοχή. Δυστυχώς τα δημόσια κονδύλια δεν αρκούν. Γι' αυτό και πραγματικά κάνω μια έκκληση εδώ να ξανασκεφτείτε με ποιο καινοτόμο τρόπο μπορείτε να μας στηρίξετε. Πώς οι άνθρωποι ζουν και τον οποίων η επιβίωση εξαρτάται από αυτήν την δραστηριότητα. Παράγουμε τρόφιμα που επίσης είναι σημαντικά για την ε, επιβίωση όλης της ανθρωπότητας. Στέφαν. Για την ερώτηση που θέσατε, να σας πω πρώτα πρώτα ότι μίλησα για την απαξίωση της ε, γης. Όχι, όχι υποτίμηση. Απαξίωση από πλευράς φύσης. Γιατί οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ασχολούνται περισσότερο με τη γη και προσαρμόζονται περισσότερο καλύτερα ε, και στα ε, μέτρα για το περιβάλλον, τα οικολογικά. Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις όχι. Όπως σας είπα, είμαι αντιπρόεδρος ε, της οργάνωσης των καλλιεργητών, των, των μικρών καλλιεργητών. Αλλά έχουμε και μεγάλες εκμεταλλεύσεις στην οργάνωσή μας. Έχουμε από 30 εκτάρια εκμεταλλεύσεις στην οργάνωσή μας μέχρι 150. Δεν ξέρω αν ε, ρωτήσατε και εμένα. Είπα για το Υπουργείο Γεωργίας ότι δεν υποστηρίζει τις μικρές εκμεταλλεύσεις. έχουμε κάποιες ενισχύσεις αναεκμετάλλευση. Δεν έχουμε αναεκμετάλλευση. Τους έχουμε διαφορετικό σύστημα στην Τσεχία. Έχουμε πληρωμές ανά εκτάριο, όχι ανά επιχείρηση. Αν έχω 20 εκτάρια στην εκμεταλλευσή μου, θα πάρω, θα πάρω 5.000 κορώνες επί 20. Και αυτό ισχύει για όλες τις εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν κάποιες με 10 ή 20.000, 30.000 ε, εκτάρια, οπότε παίρνουν την ενίσχυση επί 10.000-30.000. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα να ακούσω τις απόψεις σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση. Έχω αυτή τη μακρά πείρα όσον αφορά τις κοινωνικές εκμεταλλεύσεις. Οπότε, ξέρω ότι περί να πρόκειται γιατί ζω στην Ήπεθρο και θα συνεχίσω να ζω. Αλλά το θέμα είναι αυτό που σας είπα. Θα πρέπει η τσεχική δημοκρατία να υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Από 6 δηλαδή μέχρι 50 εκτάρια. Και έτσι θα πρέπει να έχουμε κάποιες πληρωμές αναδιανεμητικού χαρακτήρα. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει είτε με κάποιο είδους φθήνοντα χαρακτήρα των ενισχύσεων προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Μιλάμε επίσης για κάποια, για κάποια πάνω από 100.000 ευρώ και με αυτός ο φθήνο χαρακτήρα των μέτρων και μιλώ για το ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό ο χαρακτήρα τη κατάργηση δηλαδή των ενισχύσεων για τι επιχειρήσει, για τι εκμεταλλεύσει πάνω από 1500 εκτάρια, να βοηθούν οι μικρέ εκμεταλλεύσει. Ο πρόεδρο. Α, ώστε έτσι γίνονται οι ενισχύσει ανεξαρτήτω τη έκταση ε, των εκμεταλλεύσεων. Ο επόμενο. έχει το λόγο κύριε Άντεμς. τι γίνεται με το βιοαέριο. Το θέτει σε εμπορία το κράτος. Οπότε θα ήθελα οι πολιτικοί να βοηθήσουν τους γεωργούς. Πάντοτε θα υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις. Σε κάθε κράτος επικρατεί διαφορετική κατάσταση δεν μπορούμε να έχουμε την αντιμετώπιση για όλα τα κράτη-μέλη. Ούτε για όλους τους κλάδους. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια βάση δίκαιης αντιμετώπισης. Και επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διορυθμίες κάθε χώρας, οπότε η προσέγγιση να είναι αντίστοιχη για κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος σημερινή συνεδρία συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι η οικογενειακή εκμετάλλευση δεν είναι κατά ανάγκη μικρή εκμετάλλευση. Είναι πολύ διαφορετικές εκμεταλλεύσεις και στην Ευρώπη και παγκόσμια. και άλλου τύπου εκμετάλλευση έχουμε στην Ευρώπη, άλλου τύπου στην Αφρική. Η μικρή, αυτό που λέμε μικρή εκμετάλλευση μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Κάποτε μικρή ήταν η εκμετάλλευση που ήταν 2 ή 5 εκτάρια. Τώρα είναι 20. Τώρα, ε, γεωργία σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας. Ε, κρυφή ανεργία και πώς αποκρύπτει το πρόβλημα της ανεργίας η γεωργία. Η σημασία των μικρών εκμεταλλεύσεων σε στιγμές ε, και εποχές ε, οικονομικής κρίσης. Είναι ένα εργαλείο η οικογενειακή γεωργία για να καταπολεμήσει την ανεργία, για να απορροφήσει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, δυσκολία να αποφέρει κερδοφορία θα πρέπει ανάλογα με την περιφέρεια να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Οι περιφερειακές αρχές μπορούν να κάνουν πάρα πολλά για να υποστηρίξουν τις ε, εκμεταλλεύσεις αυτές, ειδικά τις μικρές. Γιατί αν οι εκμεταλλεύσεις είναι μεγάλες, πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες της αγοράς. Αλλά οι μικρές εκμεταλλεύσεις μπορούν να παίξουν και άλλο ρόλο. Επομένως θα πρέπει να προστατεύονται διπλά. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη τη δυνατότητά τους να δημιουργούν οργανώσεις για να επιβιώσουν στην αγορά. Θα πρέπει να προστατεύονται ειδικά από τις περιφερειακές αρχές, όχι μόνο από την ΚΑΠ. Για πρώτη φορά η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρόσεξε το πρόβλημα των μικρών εκμεταλλεύσεων, παρότι η προσοχή που δόθηκε δεν είναι επαρκής. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμα, αλλά νομίζω είναι η κατάλληλη ώρα για να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, στρέφομαι και προς τους προσκεκλημένους μας. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα της οικογενειακής γεωργίας, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Οι οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις πρέπει να υποστηριχθούν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες. Το μικρό είναι και ωραίο. Ειδικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ελεύθερο ανταγωνισμό, Εκεί το πανοχέτιο το έχουν είναι μεγάλες. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το αστιακό παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε και άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε. Ευχαριστώ την κυρία Κιώστιγκερ από την Αυστρία. Πρέπει να είναι περήφανη για το παράδειγμα που δίνει. Αλλά βλέπουμε ότι και στα νέα κράτη-μέλη αλλάζει η γεωργία ε, μετά την εποχή του κομμουνισμού. Καταληκτικά σας ευχαριστώ όλους. Ήταν πολύ καλή αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το λάβει υπόψη και το νέο κοινοβούλιο που θα μας έρθει μετά τις εκλογές. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει σε 7 Απριλίου. Θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολη αυτή η συνεδρίαση με πολλά θέματα, όπως ήταν δύσκολη και η σημερινή πρωινή συνεδρίαση, λόγω των αποφάσεων που ετοιμάζουμε για τις κατεξιοδότηση πράξεις. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς και εμείς σας ευχαριστούμε για τον επιπλέον χρόνο τους. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, κλείνω εδώ τη συνεδρίαση. Ελπίζω να ανακτήσει την υγεία του ο πρόεδρος, να γίνει καλά. Αυτά κλείνουμε εδώ. Γεια σας. Thank you. Thank you. Thank you.